<laughs> Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής.